Περνούμε στο επόμενο θέμα. Ιράκ. Απαγωγές και κακοποίηση γυναικών. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους, αλλά σας παρακαλώ να σέβεστε απολύτως το χρόνο σας. είμαι υποχρεωμένος να σας διακόπτω. Μόλις τελειώνει ο χρόνος σας. Νομίζω ότι είναι φυσικό και επόμενο. Έχουμε πάνω από 18 ομιλητές. Ο κύριος Κάμπελ, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως πρόεδρος ε, της ε, αποστολής για τις, ε, της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις μας με το Ιράκ θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξη της αντιπροσωπείας μας για να βοηθήσουμε το Ιράκ να δημιουργήσει μια πιο δίκαιη κοινωνία που να προστατεύει τα δικαιώματα των γυναικών. Καταδικάζω τις ε, ε, βαρβαρικές, τις βάρβαρες δολοφονίες ε, των πολεμιστών του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ. Τέτοιες πράξεις αποτελούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Από το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος έχουν διαπραχθεί αυτές οι πράξεις οι οποίες είναι απάνθρωπες είναι εις βάρος ε, μελών ε, των ε, θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων όπως είναι η Κουρδική, η Τουρκμανική και άλλες. Εξαναγκάζονται να αλλαξοπιστήσουν και έχουμε εγκλήματα βιασμού και άλλα και ένα λεπτό είπαμε λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Καστάλντο για ένα λεπτό αυστηρά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ΙΖΙΣ έχει δημιουργήσει φέτος ένα σύστημα συστηματικής παραβίασης, ένα είδος συστηματικής παραβίασης κάθε ανθρώπινο δικαιώματος. Αυτές οι φροκαλαιότητες είναι όργανο προπαγάνδας στα χέρια των ανθρώπων αυτό. 11.000 ε, γυναίκες είναι σκλάβες ε, με προορισμό να γίνουν ε, σεξουαλικές σκλάβες εδώ βλέπουμε τι έχει γίνει σε, πόλεις όπως, σε περιοχές όπως η Μοσούλη και βλέπουμε να μην υπάρχει έλεος ούτε για ε, μικρά κορίτσια. Τι κόσμος είναι αυτός που αυτά τα σεξουαλικά εγκλήματα είναι καθημερινότητα στις περιοχές αυτές. Ξέρουμε ότι η διεθνή κοινότητα έχει επιβάλει ένα απαγορευτικό όριο για τα πυρηνικά όπλα ή τα χημικά. Όμως εδώ βλέπουμε ένα πιο καταστρεπτικό όπλο, ε, τη σεξουαλική βία που είναι ένα όπλο που μπορεί να καταστρέψει την ίδια την ψυχή ενός ανθρώπινου όντως. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιώντας και χρηματοδοτώντας ανθρώπους που μπορεί να το χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή βίας ως όπλο είμαστε όλοι ένοχοι. Ένοχοι γιατί παραμένουμε στα λόγια. Ευχαριστώ. Κύριος Άλαν Σμιθ για ένα λεπτό απολύτως αυστηρά. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Στο λεπτό που μου δίνετε θα κάνω ό,τι μπορώ για να παρουσιάσω την ε, τρομακτική κατάσταση στο Ιράκ. Ε, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η επέμβαση στο Ιράκ ήταν ε, καταστροφική αποτυχία πολιτικής της δυτικής κοινωνίας και θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Έχουμε ρίξει στην Άβυσο στο Ιράκ, υποφέρουν οι γυναίκες, οι άντρες και τα παιδιά και είναι σημαντικό ότι με το ψήφισμα αυτό εξετάζουμε την κατάσταση των γυναικών. Υπάρχουν πολλά θετικά σημεία στο κείμενο, ιδιαίτερα το σημείο 12 αναφέρεται στην κοινωνία των ατόμων ε, ΛΟΑΔ. Ε, επίσης αναφερόμαστε ε, στο ψήφισμα του ΟΗΕ 1325. Υπάρχουν κάποιες ιδέες για το πώς θα βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων αυτών. Έχουμε όμως ιστορική ευθύνη απέναντι στους άντρες, τις γυναίκες και τα παιδιά του Ιράκ να μην τους εγκαταλείψουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ιώζεφ Βάιντενχολτ. Για 1,5 λεπτό. Ακούμε από το βόρειο Ιράκ χιλιάδες γυναίκες και παιδιά σε καταβλισμούς πώς ζουν. Αισθανόμαστε ότι έχουμε γυρίσει στο μεσαίωνα, σαν να μην υπήρχε ποτέ ε, η σύμβαση της Χάγης ή ε, θεμελιώδης χάρτης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι εξτρεμιστές, ε, παράφρονες καταργούν οτιδήποτε έχει πετύχει μια προοδευτική κοινωνία. Οι Γεζιντοί υφίστανται τρομερές ε, κατάφορες παραβιάσεις των δικαιωμάτων, κυρίως τα κορίτσια και οι γυναίκες. Ε, ταπεινώνονται, υφίσταται σεξουαλική κακοποίηση, τους στερούν την ε, προσωπική τους ακεραιότητα, τις πουλάνε δούλες στα σκλαβοπάζαρα. Δεν μπορούμε να τα δεχόμαστε αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό θέσαμε και αυτό το αίτημα για τα κατεπήγοντα και ελπίζουμε να μπορέσουμε και εμείς να συνεισφέρουμε. Η ε, δημόσια διεθνής κοινότητα να ασχοληθεί με αυτή τη βαρβαρότητα και να τερματίσει επιτέλους αυτές τις καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζεράρ Ντεπρέ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, συνάδελφοι, μέσα σε δύο μέρες έχουμε δει δύο από τα βασικά σημεία θρικαλαιοτήτων για την ανθρωπότητα σε αυτήν την φάση. Χθε ο, ο, ο δόκτωρα Μουκουέγγε μα μίλησε για την κατάσταση των γυναικών στην ε, Δημοκρατία του Κονγκό. Σήμερα βλέπουμε τι βίε πράξει κατά γυναικών και παιδιών στο Ιράκ και δεν μπορούμε παρά να πούμε ότι είναι ανπαράδεκτο όλα αυτά. Σεξουαλική βία, βιασμοί, απαγωγές, ε, κακοποίηση κατά γυναικών και παιδιών και πώληση σε σκλαβοπάζαρα των γεζιτών γυναικών και παιδιών στη Μοσούλη. Καταδικάζουμε λοιπόν έντονα αυτέ τι επιθέσει και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν την τραγική κατάσταση παιδιών και γυναικών στο Ιράκ και τη Συρία. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που για μένα είναι το σημαντικότερο είναι ότι ζητούμε και ολοκληρώνω από την κυβέρνηση του Ιράκ να εγκρίνει το καθεστώς του Διεθνούς Δικαστηρίου για να ε, καταδικάσει τα εγκλήματα πολέμου στο Ιράκ. Ευχαριστούμε κύριο Περμοή, για ένα λεπτό. Ε, Είναι σκέτος εφιάλτης, γολγοθάς αυτό που ζουν οι γυναίκες. Ε, σε αυτό το φάντασμα κράτος, υποτίθεται ε, το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος, που προέκυψε από τη διάλυση του Ιράκ και τη Συρία. Το 2004, τι είπαμε, το 1959 ε, μετά την ε, λαϊκή κοσμική επανάσταση είχε προκύψει ένας ε, κώδικας που έδινε στις γυναίκες πολλά δικαιώματα και αυτά τα κατήργησε η Συμμαχία το 2004 και το υπεκατέστησε από ένα άλλο κώδικα που δίνει εξουσία στους φιλάρχους και στους ε, θρησκευτικού ηγέτες να ορίζουν τις μοίρες των γυναικών. Και όχι μόνο το ISIS και η Ιρακινή κυβέρνηση, η στρατιωτικές εταιρείες, υπηρεσίες ασφαλείας, πολυεθνικές, οι πάντες ε, κάνουν διακρίσεις κατά των γυναικών και ή των ΛΟΑΔ έχοντας καταργήσει τον πιο προοδευτικό κώδικα που ίσχυε στο παρελθόν. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να τηρήσουμε στάση αποχή σε αυτό το ψήφισμα. Κύριο κύριος Κέλαμ για ένα λεπτό. Οι γυναίκες έχουν γίνει πεδίο μάχης και ε, μέσα πολέμου. Και στο Ιράκ οι Ισλαμιστές ε, τρομοκράτες έχουν δημιουργήσει μια ανθρωπιστική κρίση, έχουν εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδους ανθρώπους ε, και από τον τον Οκτώβριο ε, μεταξύ 5 ε, και 8.000 γυναικών ε, κρατούνταν ως σκλάβες, δείχνουν στοιχεία του ΟΗΕ. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση και να καταδικάσει την μεταχείριση των γυναικών στο Ιράκ. Ειδικοί μηχανισμοί για να βοηθήσουμε τις τραυματισμένες γυναίκες και ιδιαίτερα τις γυναίκες Γεζιτή μαζί με την ε, παροχή ψυχολογικής ε, και ιατρικής βοήθειας ε, είναι απαραίτητη. Και τέλος, θα πρέπει να επικροτήσουμε την πρόθεση της διεθνούς κοινότητας να καταπολεμήσει το Ισλαμικό κράτος. Ευχαριστώ κύριος Κέλλη. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ δύσκολο να διαβάσει κανείς το ψήφισμα αυτό χωρίς να νιώσει αποτροπιασμό. Τον 21ο αιώνα ε, έχουμε ψυχολογικές και σωματικές επιθέσεις, ε, ε, σκλαβιά των γυναικών, γυναίκες και κορίτσια πολλούνται και επίσης καταδικάζονται σε θάνατο με αμφίβολους τρόπους. Όταν ξεπερνάμε τις κόκκινε γραμμές όπως ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος επέμβαση για να σώσουμε τις ε, γυναίκες και την αξιοπρέπειά τους. Ε, και Επίσης μας απασχολούν οι ανάγκες τώρα τον χειμώνα για τους ανθρώπους τους εκτοπισμένους. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. 57 δευτερόλεπτα μίλησε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρτά Εντουάρτου. Ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση που ζουν οι γυναίκε στο Ιράκ, στο αυτό ανακηρυχθέν ε, Ισλαμικό κράτο, είναι δραματική. Πρέπει να αναλάβει έντονη δράση το Κοινοβούλιο, διότι υπάρχει σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι γυναίκε, καταναγκαστικού γάμου, βιασμού, δουλεία, ε, πώληση στην αγορά τη Μοσούλη, είναι καταστάσει που τι ζουν καθημερινά. Εδώ λοιπόν ε, ξέρουμε ότι πριν από 15 χρόνια τα πράγματα ήταν τελείω διαφορετικά. 15.000 γυναίκε για ζήτησε θεωρούνται ε, αγνοούνται αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι στο Ιράκ υπάρχουν, ε, υπάρχει βία για λόγους θρησκευτικού και ε, εθνοτικούς. Αλλά δεν είναι μόνο η θρησκεία ο λόγος. Οι γυναίκες είναι τα πρώτα θύματα του πολέμου και έχουν γίνει ένα νόμισμα ε, που χρησιμοποιείται ως όπλο. Εδώ λοιπόν το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει αυτό το ψήφισμα για να αποστείλει ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους. Το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον την τη Αρμοστία του. Και θα ήθελα να πω λίγα λόγια και για την κατάσταση στην Ευρώπη. Ο κύριος Τσανέσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Να μην μιλάμε πλέον ε, κάστρα στην άμμο με τα λόγια μας, διότι βλέπουμε ότι αυτά τα έχει γκρεμίσει επανειλημμένο στο Ισλαμικό κράτος με τις πράξεις του. Υπάρχουν σοβαρά σφάλματα που έχουν διπραχθεί από τις ε, Ιρακινές αρχές και εμάς ε, στη Δύση. η παθητική και η παθητική στάση, η αδράνεια των Ιρακινών αρχών δείχνει κάτι. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε γιατί αυτή η εξάπλωση του, Ιρα... του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ και τη Συρία. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα από ότι να διαμαρτυρόμαστε με τα λόγια. Θα πρέπει να αναλάβουμε δράση ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αυτό που τώρα συμβαίνει μας θυμίζει καταστάσεις του Μεσαίωνα και του 21ου αιώνα θα πρέπει να πιέσουμε το Συμβούλιο και να αναλάβει αποφασιστική δράση σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστούμε κυρία Σακοράφα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κάτι πριν ξεκινήσει ο χρόνο, μου θα σα παρακαλέσω να μου διαθέσετε το ένα λεπτό και δέκα δευτερόλεπτα όπω σε όλου του συναδέλφου, ακριβώ γιατί δεν υπάρχουν δύο ταχυτήτων συνάδελφοι μέσα σε αυτήν την αίθουσα. Σα παρακαλώ πολύ. Κύριοι συνάδελφοι, πειθαρχήστε μου παρακαλώ το χρόνο. Το χρόνο μου κύριε Πρόεδρε είστε μου σας παρακαλώ το χρόνο. Κύριοι συνάδελφοι, με πέντε μήνες σε αυτό το κοινοβούλιο και σε αυτό το διάστημα έχουμε εκδώσει ψηφίσματα που καταδικάζουν τη βία και τις δολοφονίες αμάχων παιδιών, γυναικών, θρησκευτικών μειονοτήτων. Ψηφίσματα που καταδικάζουν μόνο τα αποτελέσματα και όχι τα αίτια και τις πολιτικές που τα προκαλούν. Το σημερινό αναφέρεται στο Ιράκ. Κύριοι συνάδελφοι, το βοβαρθήσαμε, κάναμε εισβολή, το διαλύσαμε και τώρα ζητάμε από το χάος που δημιουργήσαμε να σεβαστεί ανθρώπινες ζωές και δικαιώματα και θα φύγουμε με ήσυχη τη συνείδησή μας ότι επιτελέσαμε το καθήκον μας. μόνο όταν αποφασίσουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους ένα λίτρο πετρέλαιο πόσες ζωές μια ουγγιά χρυσού πόσες ζωές ένα κυβικό αέριο πόσες ζωές μια μονάδα στο χρηματιστήριο πόσες ζωές μόνο όταν απαντήσουμε σε αυτά με ειλικρίνεια τότε ίσως να αξίζει να ελπίζουν σε εμάς οι γυναίκες και ο λαός του Ιράκ, της Συρίας, της Παλαιστίνης, του Αφγανιστάν, της Λιβύης και της Ουκρανίας. Κύριοι συνάδελφοι, είναι μεγάλος ο κατάλογος και θα μεγαλώνει όσο συνεχίζουμε να νιώθουμε μικροί και να συμπεριφερόμαστε ανάλογα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Χτες ακούσαμε το δόκτωρα Μοκβέγε ε, περιγραφές πάρα πολύ εύγλωτες ε, για τα όσα συμβαίνουν στο Κογκό στη σεξουαλική κατοικοποίηση. Τόνισε συνεχώς ότι είναι όπλο πολέμου αυτός ο βιασμός σε καιρό πολέμου και μεθοδικά γίνεται. Και σήμερα βλέπουμε ένα άλλο πόλεμο που ακριβώς ε, αποσκοπεί στη καταστροφή των γυναικών και των κοριτσιών και στην ταπείνωσή τους. Από το Σεπτέμβριο τα ακούμε αυτά, ιδιαίτερα κατά των οικογενειών οι γυναίκες και τα κορίτσια ξεχωρίζονται από τις οικογένειές τους, αναγκάζονται, σε γάμους με πολεμιστές του ISIS και τους πουλάνε και στα σκλαβοπάζαρα. Αυτή η βία κατά των γυναικών είναι τμήμα της στρατηγικής του ISIS και γενικότερα της ομής και σκεάς προσπάθειας να σβηστεί ε, κάθε ίχνο ζωής που δεν είναι Άραβας ή μουσουλμάνος στην περιοχή. Ε, θα πρέπει ε, να σκεφτούμε δικαστικές ενέργειες κατά των ξένων μαχητών ε, στην Ευρώπη. Αλλά αυτά δεν αρκούν. Γι' αυτό ε, απαιτούμε από την η Ιρακινή κυβέρνηση να κυρώσει το καθεστώς της Ρώμης ο πρόεδρος διακόπτει την Ολομέλεια. Κοράω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση τη Διεθνού Αμνηστία, στο Ιράκ υπάρχει προσπάθεια εθνοκάθαρση στα βόρεια τη χώρα. Εκατοντάδε, για να μην πω χιλιάδε, ε, γυναίκε και παιδιά των γεζιτών ε, είναι αγνοούμενοι. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι έχουν υποπληθεί σε σοβαρά και φρικτά βασανιστήρια. Υπάρχει προσελητισμό, υπάρχει βία, ε, αλλά στι γυναίκε τα πράγματα είναι χειρότερα. Παλακίδε, ερωτική γάμη, σεξουαλική βία από τα τεύματα που επιτίθενται. Με πολλές φορές στόχο την ε, ίδια τη δολοφονία τους. Ε, εδώ λοιπόν δεν ξέρουμε τον αριθμό των θυμάτων. Οι γυναίκες αυτές δεν μπορούν να περάσουν τα σύνορα της χώρας ε, και τις περιοχές που ελέγχει το Ισλαμικό κράτος. Υπάρχουν σοβαρότατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ που μπορούν να θεωρηθούν είτε εγκλήματα πολέμου είτε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. δεν μπορούμε όμως να παραμένουμε αδρανείς. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να παρέμβουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ε, ευχαριστώ κύριο Φερόν για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ιράκ σήμερα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων και όλη η ευθύνη πολλών από εσά και από του φίλου σα. Πριν από 25 χρόνια ο Τζορτ Μπρούς, εν ονόματι του πετρελαίου, ε, ε, έλαβε την ολέθρια απόφαση να κάνει μια ανεπανάληπτη επιδρομή σε μια χώρα ενωμένη, κοσμική, που σεβόταν τι μειονότητες οι περισσότεροι ε, από το λαό του Ιράκ συμφωνούσαν με αυτό το κράτος που είναι μια χώρα με πανάρχια παράδοση και ιστορία. Συμπέρασμα ε, και συνέπεια ε, είναι τώρα βορρά στα χέρια της χειρότερης ιδεολογίας που υπήρξε ποτέ. Σκανδαλώδης ήταν η επιχείρηση του 2003, αυτή τη φορά από το νεότερο, τον Ιόπους. Ε, και έχουμε ε, το ISIS ε, χάρη στην αμερικανική πολιτική που του στήριξε ανοιχτά και καλυμμένα και με την τουρκική συνενοχή. Εξακολουθείτε όμως να θέλετε να υποστηρίζετε Ισλαμικές ιδεολογίες ομάδας παντού στην περιοχή. Ο Πρόεδρος Διακόπτω τον ομιλητή, τελείωσε ο χρόνος σας. Η κυρία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, είμαστε μάρτυρες μιας από τις πλέον βίες επιθέσεις ε, από το Ισλαμικό κράτος κατά των γυναικών με βιασμούς, δολοφονίες, με μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Κορίτσια και γυναίκες ε, πέφτουν θύματα ε, βίες μεταχείρισης σαν να είναι εμπορεύματα και μιλάμε για διακρατικέ διαστάσει αυτού του φαινομένου, διότι ξεπερνά τα σύνορα ενό κράτου το Ισλαμικό κράτο. Το λεγόμενο, αυτοποκαλούμενο Ισλαμικό κράτο. Πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε δρυμία κριτική και να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή σεξουαλική βία και αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα κατά των γυναικών. Όπω είπε ένα συνάδελφο, ο βιασμό είναι ένα τρομερό όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταστρέψει μια ανθρώπινη ψυχή. Πρέπει να τυπονίσουμε λοιπόν του υπευθύνου. Και να απευθύνουμε έκκληση στις Ιρακινές αρχές για να εγκρίνουν και να αποδώσουν τους υπευθύνους στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ευχαριστούμε κύριος Μπέλντερ για να... Ε, κύριε Πίτροπε, είναι ε, τρομερά τα δεινά των γυναικών στο Ιράκ. Θέλω να σας ρωτήσω τα εξής. Υπάρχουν προγράμματα βοήθειας, ψυχολογικής υποστήριξης για αμέτρητες γυναίκες και κορίτσια που βιάζονται. περίπου 2 εκατομμύρια ε, είναι οι χείρες που τις ε, παντρεύουμε το στανιό είτε με τη μούτα που είναι ένας ε, γάμος προσωρινός είτε οριστικά ή με πολυγαμία. Επίσης δεν υπάρχει ελάχιστο όριο ηλικίας για τους γάμους. Έχουμε ρυθμίσεις για κορίτσια μέχρι 9 ετών που ζητούν διαζύγιο. Τι θα γίνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει καμία δράση απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βεργία, για ένα λεπτό. Το ψήφισμα αυτό θεωρητικά αφορά τις απαγωγές και την κακομεταχείριση των γυναικών στο Ιράκ. Όμως, όταν, τα θύματα πέφτουν, ε, όταν οι γυναίκες πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης ε, οπουδήποτε από τρομακρατικές ομάδες που σπήρουν τον τρόμο παντού, τι κάνουμε, ε, βιασμοί, καταναγκαστική γάμη, προσελητισμός, πώληση των γυναικών, στο όνομα της θρησκείας. Οι χριστιανοί και οι είναι τα πρώτα θύματα αυτών των δύο ενεργειών. Όσο πιο νεαρές είναι οι συνθήκες τόσο ακριβότερες είναι στην αγορά. Ε, με το ψήφισμα αυτό όμως η δράση μας είναι πολύ αδύναμη. Διότι πρέπει να μιλ... δεν μπορούμε απλώς να μιλάμε γενικόλογα για την κατάσταση στο Ιράκ. Ε, μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουμε τώρα την αντίδρασή τους αν έχουν αφήνει για την αποδιοργάνωση της χώρας αυτής. Το ξαναλέω λοιπόν, ο τρόπος που τα κατεπήγοντα τα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα τα αντιμετωπίζουμε σε αυτό το εμικύκλιο γίνεται αναποτελεσματικός και ακατανόητος. Δεν είμαστε αποτελεσματικοί. Όλα αυτά που είπατε δεν ε, κάνουν κάτι για την ουσία. Ευχαριστούμε κυρία Τζούλια Μόη για ένα λεπτό. Πρόεδρε, στις 25 Νοεμβρίου γιορτάσαμε την Διεθνή ημέρα για την ε, απάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Όμως αυτός ο εορτασμός είναι κενός νοήματος, βλέποντας τι συμβαίνει στο Ιράκ εξαιτίας των τρομοκρατών του Ισλαμικού κράτους. Οι γυναίκες των γεστών ε, πρέπει κάθε μέρα να ζουν βίες μορφές αντιμετώπισης με, κατα... με βιασμούς, σεξουαλική δία, προσαλ... προσελητισμούς, συνοπτικές εκτελέσεις, πώληση σε σκλαβοπάζαρα. Καταδικάζουμε αυτές τις ενέργειες και ζητούμε από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψουν ειδικά μέτρα για να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα αυτών των γυναικών. Ελπίζω επιπλέον η κυβέρνηση του Ιράκ να γίνει σύντομα μέλο του Διεθνού Δικαστηρίου τη Χάγη, εγκρίνοντά το, προκειμένου να επιτρέψει την δίωξη των ε, υπευθύνων για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα ε, που έχουν διαπραχθεί από το Ισλαμικό κράτο. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ όσοι τώρα στην αίθουσα να καθίσουν όσο το δυνατόν ησυχότερα, διότι θα πρέπει να ακούσουμε τον Επίτροπο Στυλιανίδη, ο οποίο θα κλείσει τη συζήτηση αυτή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα και να εκπροσωπώ την ε, Αντιπρόεδρο Φεντερίκα Μοκερίνη για να συζητήσουμε ένα θέμα που μας ανησυχεί πολύ. Ε, μας ε, δυσαρεστούν ε, όπως και όλους εσάς οι καθημερινές αναφορές βιοπραγιών εις βάρος γυναικών και κοριτσιών. Έχουμε ακούσει απαγωγές, αναγκαστικούς γάμους, σκλαβιά, σεξουαλική κακοποίηση και ότι τις αναγκάζουν να αλλαξοπιστήσουν τις γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες. με την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει καταδικάσει τις βάρβαρες αυτές πράξεις και έχει ζητήσει να αποδοθούν ευθύνες ε, σε όσους έχουν διαπράξει αυτά τα εγκλήματα. Ε, και έχουμε ε, υποβάλει έτοιμα στον ε, αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε ζητήσει να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με την παραβίαση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Πρόεδρος, ε, κύριε Επίτροπε, θα ξαναζητήσω από όλους να καθίσουν ε, ήσυχα για να ακούσουμε τον Επίτροπο και να κλείσουμε τη συζήτηση. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Η Ιρακική κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει την, την έρευνα πάνω σε όλες τις υποθέσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβίαση του κράτους δικαίου. Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει αναθεώρηση του ποινικού συστήματος και να δημιουργηθεί μια κουλτούρα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα πρέπει να διασφαλιστεί η ισότητα όλων των πολιτών απέναντι στον νόμο. Αυτό θα ε, αποτελέσει σημαντικό στοιχείο της ε, διαδικασίας ε, συμφιλίωσης. Πολλές από αυτές τις πράξεις που διαπράττονται στο Ιράκ αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γι' αυτό Ζητάμε το Ιράκ να δεχθεί τουλάχιστον τη δικαιοδοσία του ε, Διεθνούς ε, Ποινικού Δικαστηρίου ε, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Ρώμης. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί το κράτος δικαίου και η σωστή κυβέρνηση στο Ιράκ. Νέο πρόγραμμα ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ ξεκίνησε αρχές Σεπτεμβρίου. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μια σειρά προγραμμάτων βοήθειας που συνδέονται ε, πιο άμεσα με την προστασία γυναικών και παιδιών συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος ε, που να καθορίζει μια στρατηγική για την προστασία των γυναικών και βοήθεια ε, στα θύματα ε, Σεξουαλική ε, βία ε, και εμπορία ανθρώπων. Η προστασία ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τεράστιος ο αριθμός προσφύγων και η Ευρώπη έχει αυξήσει τις, τις ανθρωπιστικές της δράσεις. Θα, απο... θα απαιτηθεί λοιπόν βοήθεια προ τα θύματα όλων των ειδών βία, συμπεριλαμβανομένη τη σεξουαλικής. Να κλείσω τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει την κυβέρνηση του Ιράκ στου δύσκολου αυτούς καιρούς και θα αυξήσει τις προσπάθειες για να ανακουφίσει ε, τις συνθήκες των ε, θυμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ε, έχω λάβει 7 προτάσεις ψηφίσματος. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αμέσως στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.